Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας σαν υποεπιτροπή άμυνας. Να σας πληροφορείτε ότι κάποιες γλώσσες δεν υπάρχουν όπως τα δανέζικα, τα φιλανδικά και τα μαλτέζικα. Είναι η τελευταία συνεδρίαση φυσικά εφέτος, η τελευταία συνεδρίαση με τη Σουηδική Προεδρία και αν δεν έχετε αντιρρήσεις με την ημερήσια διάταξη θεωρείτε δεκτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα θέλαμε να καλωσορίζουμε τον κύριο Λοφσκούκ, Σουηδό πρέσβη, προεδρεύοντα το PSC, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα επιτεύγματα της Σουηδικής Προεδρίας στον τομέα της κοινή πολιτικής ασφάλειας, όπως ονομάζεται στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πρέσβη, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω εξ ονόματος της Υποεπίτροπης για το σωστό πνεύμα συνεργασίας το οποίο κυριάρχησε κατά τη διάρκεια αυτής της εξάμενης περίοδου. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, κάτι το οποίο θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες δυνατότητες δράσης. Στις 8 Δεκεμβρίου του 2009, μια συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων έγινε στις Βρυξέλλες, σχετικά με την επιχείρηση Άλτεα στην Βοσνία ερζιγομβίνη και την επιχείρηση Αταλάντα στην ακτή της Ομαλίας και ο κύριος πρέσβης Κόγκ θα σχολιάσει τις δύο αυτές εξωτερικές δράσεις. Υπάρχει επίσης και μια πιθανή αποστολή για την ενίσχυση και εκπαίδευση μάλλον των σομαλικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο θα συνεισφέρει στην αποκατάσταση της τάξης στην Σομαλία. Και η κυρία Άστον, η Βαρόνη Άστον θα είναι παρούσα σε μία από τις μελλοντικές μας συναντήσεις, όπως επίσης και κάποιος εκπρόσωπος της Ισπανικής Προεδρίας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και δίνω στον πρέσβη Σκόκ το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε για τη Σουηδική Προεδρία. και εμείς από πλευράς μας έχουμε εκτιμήσει ιδιαίτερα τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με τις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. και σας ευχαριστώ που παραμείνατε εδώ μετά από τη στρατηγική παρουσίαση που έκανε ο Κάρλ Μπίλτ και αυτοί που έχετε μείνει υποθέτω ότι είστε εμπειρογνώμονες της κοινή πολιτικής άμυνας. Θα σας πω ότι προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και να αναφερθώ στην πιθανή αποστολή στην Σομαλία, κάτι το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Ξεκινώντας να πω ότι όταν ήμουν εδώ την τελευταία φορά, στις 7 Σεπτεμβρίου δηλαδή, είχα εκθέσει κάποιες από τις, προεδρι... από τις προτεραιότητες της Προεδρίας και νομίζω ότι έγιναν γενικότερα ευνοϊκά δεκτές από την πλειοψηφία της Επιτροπής σας. Και σήμερα θα προσπαθήσω να σας δώσω μια καλύτερη ενημέρωση λίγο πριν κλείσουμε αν θέλετε τα βιβλία απολογισμού της Σουηδικής Προεδρίας. Νομίζω ότι από πλευράς μας ε, μπορούμε να είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Όπως έχετε παρατηρήσει και από την παρουσίασή μου ή θα παρατηρήσετε από την παρουσίασή μου, εμείς δεν είχαμε φιλοδοξία να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, νέες περίφημες ε, πρωτοβουλίες, αλλά να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα και στο επίπεδο το πολιτικό και στο επίπεδο το στρατιωτικό και να προσπαθήσουμε αυτά να τα καλύψουμε και να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και όχι προς κάτι το ιδιαίτερα φιλόδοξο ή και εφήμερο. Ιδιαίτερα σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλειών θα έλεγα ξεκινήσαμε μια διαδικασία ελέγχου φιλόδοξη αρκετά για να καλύψουμε τα περισσότερα κενά τα οποία παρεμποδίζουν τις αποστολές μας και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και στο μέλλον. Το κάναμε αυτό σε στενή συνεργασία και με τα θεσμικά όργανα και με τα κράτη-μέλη. Στον στρατιωτικό τομέα προωθήσαμε τους τέσσερους βασικούς στόχους τους οποίους είχαμε θέσει στην αρχή της Προεδρίας και για μας αλλά και για την Ένωση και νομίζω ότι και εκεί έγιναν κάποια αρκετά σημαντικά βήματα προόδου στα οποία θα επανέλθω σύντομα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας είναι η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Όπως το είπε και ο κύριος Μαυρονικόλας, είδαμε το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και αυτό που έχει σημασία θα έλεγα είναι ότι η Σουηδική Προεδρία έτσι όπως εμείς ε, την διαχειριστήκαμε είναι το τέλος μιας εποχής σε επίπεδο κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Τα πράγματα αλλάζουν από εδώ και πέρα και ο κύριος Κάρλ Μπίλτ είπε προηγουμένως με καλύτερο τρόπο ότι έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με πιο συντονισμένο τρόπο. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από την αποστολή την οποία θα αναλάβει πλέον ο ύπατος εκπρόσωπος ή ύπατος μάλλον για τις εξωτερικές υποθέσεις. Και φυσικά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να ορίσουμε σωστά τι, τι φιλοδοξίες έχουμε από το μέλλον. Για την, υπηρεσία εξωτερικών, για την εξωτερική υπηρεσία μάλλον και αυτό θα είναι ένα νέο πεδίο στο οποίο θα πρέπει να δράσουμε σωστά για να επηρεάσουμε θετικά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον τομέα της πολιτικής ασφαλείας δεν μπορεί να λειτουργήσει η πολιτική ασφαλεία αν δεν την υποστηρίξουμε όλοι. Δηλαδή η αίσθηση της συλλογική ιδιοκτησίας των πολιτικών αυτών από την εκλογική περιφέρεια μέχρι το υψηλό εθνικό επίπεδο είναι ξεκάθαρο για να προχωρήσουμε σε σωστές πολιτικές δράσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα μπορούμε να αφήσουμε μόνο στη φροντίδα του υπάτου εκπροσώπου εξωτερικών θεμάτων. Το θέμα είναι συνολικά να νιώσουμε υπεύθυνοι όλα τα θεσμικά όργανα για τις δράσεις αυτές. Να επανέλθω όμως τώρα, μου επιτρέψτε, στα της Σουηδικής Προεδρίας για να σας μεταφέρω κάποια από τα κεντρικά στοιχεία των επιτευγμάτων μας. Να ξεκινήσω με το πολιτικό κομμάτι και να περάσω πετά στο στρατιωτικό κομμάτι και ίσως μετά να αναφερθώ και σε κάποια μεικτά θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα τελειώσω με τις ε, δράσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και την πιθανότητα της νέας αυτής εκπαιδευτικής δράσης ή δράσης κατάρτισης των ενόπλων δυνάμεων της Σομαλίας. Λοιπόν, για τις κατευθυντήριες γραμμές συμφωνήσαμε στο παρελθόν και με την Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη τις προτεραιότητές μας και τα επίπεδα φιλοδοξίας τα οποία είχαμε και αυτό μας επέτρεψε να πετύχουμε νομίζω αρκετά καλά αποτελέσματα. Το θέμα της γρήγορης ανταπόκρισης, η γρήγορης απάντησης σαν παράδειγμα. Προς την κατεύθυνση αυτή πήραμε μία απόφαση για την αναθεώρηση του CRT, δηλαδή ε, των πολιτικών ομάδων ανταπόκρισης μέσω ακριβώς των δυνατοτήτων που παρέχουν οι διάφορες χώρες, διευρύνοντας τα πεδία εμπειρογνωμοσύνης και καθιστώντας ε, την ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών πολιτικών, επαναλαμβάνω, πιο ε, ευέλικτη δηλαδή το θέμα του καθορισμού του προσωπικού που θα διαθέτουν τα κράτη-μέλη σε επίπεδο αστυνομικό, δικαστικό, ιατροδικαστικό ή ιατρικό, έτσι ώστε να αποστέλλονται σε αποστολές έρευνας αν αυτό απαιτείται. Προωθήσαμε επίσης και μία απόφαση σχετική με την προσπάθεια αποθήκευσης του υλικού, το οποίο θα πρέπει να είναι μονίμως διαθέσιμο, άμεσα διαθέσιμο θα έλεγα, και επίσης ε, το υλικό το οποίο προέρχεται από αποστολές ε, που έχουν ολοκληρωθεί να φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου στο μέλλον. Ε, σαν παράδειγμα τέθηκε το θέμα της χρησιμοποίησης των αποθηκών της αστυνομικής δύναμης στην Βοσνία. Για την χρηματοδότηση τώρα των δυνάμεων αυτών έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά με τα ενδιάμεσα μέτρα και τις γραμμές του προϋπολογισμού που θα είναι διαθέσιμες. Αυτό οδήγησε σε μια συμφωνία έτσι ώστε τα προπαρασκευαστικά ποσά για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση των πρώτων σταδίων των δράσεών μας. Το Νοέμβριο το Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη στα θέματα αυτά να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να κάνει προτάσεις σχετικά πάντα με τις, ε, με τις ε, ταχύτατες προμήθειες τις οποίες έχουμε ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρει τρόπους ταχύτερης προμήθειας προϊόντων σε τομείς όπως ε, η υγεία, η ασφάλιση, οι τηλεπικοινωνίες, ε, όπως επίσης και τα αυτοκινούμενα οχήματα σε επίπεδο θα έλεγα ενιολογικό περισσότερο έχουμε αναφερήσει την εικόνα, την ιδέα που έχουμε για τις αστυνομικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα τελευταία 7 χρόνια εμπειρίας που έχουμε συλλέξει στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Έχουμε κάνει κοινέ προσπάθειες με τα κράτη-μέλη για να διευκολύνουμε την ανάπτυξη του πολιτικού προσωπικού. Οι προσπάθειες αυτές τις οποίες κάνουμε, τις κάνουμε κυρίως εθνικά μέσω των εθνικών στρατηγικών Κάποιες χώρες είναι πιο δραστήριες από άλλες, αλλά μέσω ακριβώς και των εμπειριών τις οποίες μοιράζουμε και των γυμνασίων και ε, τεστ τα οποία κάνουμε, νομίζω ότι όλες οι χώρες είναι σε θέση να μας παρέχουν το προσωπικό το οποίο έχουμε πράγματι ανάγκη. Και εδώ θα ήθελα να σας ζητήσω να βοηθήσετε και εσείς σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε όταν χρειαστεί να καλύψουμε ε, τις ανάγκες τις οποίες έχουμε στις διάφορες αποστολές με το κατάλληλο προσωπικό, να μας βοηθούν γρήγορα τα κράτη-μέλη, γιατί μερικές φορές η έλλειψη πολιτικού προσωπικού είναι δραματική. Είναι πιο εύκολο να βρει κανείς το στρατιωτικό προσωπικό σε κάποιες αποστολές, στο Αφγανιστάν ή και αλλού, ε, και όχι να βρει δικαστές ή αστυνομικούς κτλ. Για την κατάρτιση τώρα έχουμε υπογραμμίσει τις διαδικασίες ε, ε, ε, εκπαίδευσης πριν την ανάπτυξη των πολιτικών δυνάμεων στα πλαίσια ενός συστήματος λογισμικού το οποίο έχουμε διαμορφώσει. Κάποιοι από τους στόχους λοιπόν τους οποίους έχουμε θέσει έχουν επιτευχθεί, απαιτείται όμως να συνεχιστεί η δουλειά σε όλους αυτούς τους τομείς. Πέρα όμως από τα, αποτελέσματα στα οποία έχουμε καταλήξει, νομίζω ότι έχουμε ορίσει το πλαίσιο κίνησής μας και για το μέλλον. Νομίζω ότι τα πράγματα ξεκινάνε ε, τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά λίγο καλύτερα προπαρασκευασμένη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσει τις οποίες έχει ο υπόλοιπος κόσμος σε σχέση με ε, την πολιτική ε, παρέμβασή μας, με τις πολιτι... μη στρατιωτικές δυνατότητες παρέμβασής μας. Τώρα για το στρατιωτικό κομμάτι, εμείς είχαμε τρεις τομείς. Καταρχάς, τους, τους, the issue of maritime surveillance uh, περιπτώσει, τις ένοπλες, ε, επίσης ε, και για το πρώτο κομμάτι, η φιλοδοξία μας για τους ευρωπαϊκούς σχηματισμούς μάχης, ε, προσπαθήσαμε να τους καταστήσουμε πιο εύχριστους και πιο ευέλικτους. Εμείς που προερχόμεθα από τη Σουηδία θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχηματισμοί μάχης δηλαδή, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκρινόμεθα σε κρίσεις όταν ξεσπούν. Μέχρι τώρα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιες από αυτές τις μονάδες, αλλά νομίζουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις γιατί δεν τους έχουμε χρησιμοποιήσει. Και παρόλα αυτά στην τελευταία κοινή συνάντηση ε, των Υπουργών ε, Άμυνας ε, καταλήξαμε σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το εύχριστο και το ευέλικτο των, ε, ε, ε, σχηματισμών αυτών. Έχουμε σύν τις άλλες και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τα κριτήρια για την δυνατότητα γενικότερα χρήσης τους. Για την ναυτική επιτήρηση. Η επιτήρηση των θάλασσών. Η Σουηδία έχει προσφέρει τη δική της εμπειρία από τη Βαλτική θάλασσα εκεί όπου η συνεργασία του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και έχει βοηθήσει πολύ και στα πλαίσια του αποτελεσμα... της αποτελεσματικότητας και του κόστους. Οι δυνατότητες αυτές έχουν εξεταστεί και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για ε, ένα οδικό χάρτη, όπως λέγεται, ε, για να καταλήξουμε στον καλύτερο τρόπο ναυτικής συνεργασίας ε, και ελέγχου των θαλασσών μέχρι το τέλος του 2010. Τώρα στο τέλος, το τρίτο τομέα κατά προτεραιότητα, η αμυντική βιομηχανία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πιο ανοιχτή και διαφανή αγορά επί τη βάση αυτού που ονομάζουμε απόλυτα δίκαιη κατανομή δυνατοτήτων θα πρέπει να καθορίσουμε τις παραμέτρους για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουμε. Τα θέματα αυτά των στρατιωτικών προμηθειών είναι περίπλοκα βέβαια όπως ξέρετε όλα, αλλά παρόλα αυτά υιοθετήσαμε μια πολιτική δούληση για να προχωρήσουμε σε μια αγορά στρατιωτικού υλικού ευρωπαϊκή διαφανή και ανοιχτή. Και ζητήσαμε επίσης και από την υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας να ασχοληθεί με το θέμα και να κάνει προτάσεις στο μέλλον. Σύντομα τώρα κάποια από τα ανάμεικτα στρατιωτικά πολιτικά θέματα, παιδεία, συνεργασίας δηλαδή του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα. Συγκεντρώσαμε την προσοχή μας στην ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συντονισμός ανάμεσα στα πολιτικά και στρατιωτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό αφορά και τις επί του εδάφους ανάπτυξη συνεργασία και την ανάπτυξη σε επίπεδο σχεδιασμού θα πρέπει να αναζητήσουμε ε, κοινέ λύσεις για την ανάπτυξη των πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων. Θα συζητηθεί το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια των νεαρινών συναντήσεων. Κάποιοι τομείς τους οποίους έχουμε ήδη την δυνατότητα ε, την επικοινωνία, αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, ε, την επιμελητία, τις αερομεταφορές, και θα πρέπει όλα αυτά τα μέσα να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από πλευράς κόστους. Σχετικά με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ε, αξιοπιστίας των παρεμβάσεών μας, λαμβάνουμε υπόψη θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προβληματική των φύλων ιδιαίτερα σχετικά με την εκπαίδευση και την προετοιμασία του προσωπικού που θα πάρει μέρος στις αποστολές. Ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν και προβληματική των φύλων. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι η συνεργασία με άλλου είδους εταίρους. Εδώ έχουμε προχωρήσει τη συνεργασία μας με την Αφροκανική Ένωση. Μια επιτροπή μας πήγε στην διάσκεψη, ε, συνεδρίαση μάλλον της Επιτροπής Ειρήνευσης ε, της ε, Αφρικανικής Ένωσης στην Άντις στην Άντισα Μπέμπα και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας μαζί τους. Όπως γνωρίζετε, σε σχέση με την πιθανή ε, εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού για τη Σομαλία, προφανώς η συνεργασία μας ε, για, με την Αφρικανική Ένωση για να πετύχει η αποστολή αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη έχει επίσης προωθηθεί στο παρελθόν και θα συνεχίσει να προωθείται από την Προεδρία μας Πήραμε την απόφαση πρόσφατα να συνεισφέρουμε ακόμα περισσότερο στον διάλογο που ονομάζεται Νέοι Ορίζοντες στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι ένα προσχέδιο εξυγχρονισμού των ειρηνευτικών δράσεων των Ηνωμένων Εθνών και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτής της προσπάθειας. Είχαμε συναντήσεις με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών όπως τον Αλάλο Λεχουά, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τις ειρηνευτικές ε, ε, αποστολέ και ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα Ηνωμένα Έθνη και να υπάρξει αμφίδρομη συνεργασία ανάμεσα στα δύο όργανα. Είχαμε επίσης σημαντικές μορφές αλληλοεπίδρασης πριν καθορίσουμε στις δικές μας στρατηγικές στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, στρατηγικές τις οποίες αναφέρθηκε ο Καλμπιλ προηγουμένως. Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία και με τον Νότις Χάιντερ τον υπεύθυνο της δράσης των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν και υπήρξε συνάντηση και με τους ε, προσώπους των ε, Υπουργείων Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το θέμα της συνεργασίας με τις στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το αντιμετωπίσαμε και περίπλοκο βέβαια, το αντιμετωπίσαμε σε πρακτικό επίπεδο επιτρέποντας να υπάρξουν περαιτέρω δυνατότητες αλληλοεπίδρασης ανάμεσα στην ΥΠΑ του εκπρόσωπο για τα εξωτερικά θέματα και το νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όπως γνωρίζετε, ο Ράσμουσεν επισκέφθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη του Συμβουλίου τον Νοέμβριο. Και εκεί υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της συνεργασίας ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία αποστολών. Πήρα μέρος και εγώ στο βορειοατλαντικό, στη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού ε, ε, Συμφώνου για να τους ενημερώσω για την εξέλιξη ε, της προσπάθειάς μας στις δράσεις Αταλάντα, γιατί σε καθημερινή βάση υπάρχει αλληλεπικοινωνία με τις στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή και πρέπει να έχουμε καλό συντονισμό μαζί τους. Τέλος, σχετικά με τα θέματα μείωσης του κόστους. Αναφέρθηκα, αν δεν κάνω λάθος, και θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά, το ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο δραστήρια και πιο συγκεντρωμένη σε προσπάθειες όπως αυτό της επιδιαιτησίας. Είναι πολύ σημαντικό αν πράγματι θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι σε σχέση με την παρουσία μας στη διεθνή σκηνή να είμαστε ικανοί και να επιμορφώσουμε το προσωπικό μας και τους πρέσβεις μας στα θέματα της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης και της επαφής με, ε, με, ε, με τρίτους εμπλεκομένους. Υπολογίζουμε την, στην υποστήριξη χωρών όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή η δημοκρατία, η δομινικανή δημοκρατία και τα λοιπά στις προσπάθειες Τουρκία βέβαια και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε μια οργάνωση η οποία να είναι ανοιχτή και να καλοδέχεται τις διάφορες χώρες οι οποίες θέλουν να συνεισφέρουν στις προσπάθειες τις οποίες αναλαμβάνουμε. Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης αυτής της αλληλεπίδρασης, όχι μόνο για να καλύψουμε τα πρακτικά κενά τα οποία διαπιστώνουμε ότι έχουμε, αλλά αν υπάρχουν περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στις δράσεις μας, αυτός είναι ένας διαφορετικός τρόπος εξαγωγή σε εισαγωγικά αν θέλετε και της εμπειρογνωμοσύνης και των αρετών και αξιών τις οποίες έχουμε και θέλουμε να προωθήσουμε σε κάθε ευκαιρία. Πριν ολοκληρώσω, και να ακούσω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας, λίγα λόγια για τις αποστολές τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας δεν έχει υπάρξει, ήμασταν τυχεροί κάποιες σοβαρές κρίσεις στις δράσεις αυτές, αν και πολλές από αυτές γίνονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και αναφέρουμε στη Γεωργία, τη Σομαλία και την Αταλάντα, η οποία είναι ενός έτους σήμερα, έχει γενέθλια και είναι αρκετά επιτυχής αλλά παρόλα αυτά είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πολιτικό και στρατιωτικό περιβάλλον. Η Βαρονιά λοιπόν συμφωνεί λέγοντας ότι θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε έτσι ώστε οι χιλιάδες ανδρών και γυναικών κάτω από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες εξωτερικές δράσεις να καλύπτονται πλήρως, να νιώθουν ότι τους φροντίζουμε, φροντίζουμε την ασφάλειά τους. Το κοσφοπέδιο έχει και εκεί μια δική μας εξωτερική δράση πολύ περίπλοκη, αλλά με τύχη κάτω από τις συνθήκες αποφύγαμε ε, σημαντικές ε, δυσκολίες, εκτός από το θέμα του βανδαλισμού, το οποίο έχουμε συζητήσει πρόσφατα. Δεύτερον, ένα γενικότερο θέμα είναι η έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού παραμένει πάντα ένα πρόβλημα. Συζητήσαμε το θέμα της αποστολής στο Αφγανιστάν προηγουμένως. Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για να στείλουμε περισσότερα αστυνομικά όργανα στο Αφγανιστάν. Έχουμε προσθέσει άνω των 100. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στους 400 του οποίους είχαμε θέσει σαν στόχο. Τρίτον, για την αποστολή εκπαίδευσης στη Σομαλία. Έγινε μια πρώτη συζήτηση στις αρχές του φθινοπόρου για μια πιθανή αποστολή. Το Συμβούλιο ξέρετε ότι συμφώνησε σε μια δράση η οποία ονομάζεται διαχείριση της κρίσης και θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό και με την Ισπανία η οποία θα είναι η υπεύθυνη χώρα για να προωθήσει αυτή την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά οι αποφάσεις τις οποίες πήραμε μέχρι τώρα δεν θίγουν σε καμία περίπτωση την δυνατότητα ανάληψης της συγκεκριμένη δράσης. Για να λειτουργήσει όμως η συγκεκριμένη δράση, και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσω αυτό, και για να πετύχουμε το στόχο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων της μεταβατικής κυβέρνησης στη Σομαλία, κάποιοι τομείς θα πρέπει να προωθηθούν και προς το παρόν αυτό δεν έχει γίνει. Θα πρέπει δηλαδή να εντάξουμε το θέμα αυτό στα γενικότερα πλαίσια της πολιτικής μας, το κέρας της Αφρικής. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επίσης και σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τους διεθνείς εταίρους και το πώς εκτιμούν την κατάσταση ασφαλείας στη Σομαλία. Θα πρέπει να το κάνουμε επίσης και σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και να κατανείμουμε την αποστολή του καθενός γιατί αυτή είναι ήδη εκεί ενώ εμείς δεν είμαστε ουσιαστικά. Και θα πρέπει να υπάρξει και ανάληψη υποχρεώσεων από πλευρά της μεταβατικής κυβέρνησης να συνεργαστούν μαζί μας και να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις όπου εκεί τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κομβικά για να τους βοηθήσουμε. Θα πρέπει να δούμε επίσης και τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς όταν εκπαιδευτούν και επιστρέψουν στη Σομαλία. Θα πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητες επιτόπου έτσι ώστε να παραμείνουν πιστοί στις μεταβατικές κυβερνήσεις και να μην προσχωρήσουν σε ε, ακραίες ομάδες. Αν δεν το πετύχουμε αυτό τότε θα προκαλέσουμε βλάβη στην προσπάθεια που γίνεται στη Σομαλία. Πάντως η συζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα δεν νομίζω με ικανοποιητικό τρόπο και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Σομαλία θα πρέπει να, θα έλεγα, να περιλαμβάνει σίγουρα μια μεγαλύτερη σταθερότητα σε επίπεδο κυβερνητικό. Αυτά κύριε Πρόεδρε, μίλησα για πάρα πολλή ώρα, περιμένω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Εμείς οι σοσιαλιστές σήμερα δεν θα εκμεταλλευτούμε την απουσία των χριστιανοδημοκρατών συναδέλφων που έχουν πάει όλοι στη Βόνη στο συνεδριό τους. Πάντως σε όλα αυτά τα θύματα έχουμε θα έλεγα συγκλίνει στο εσωτερικό αυτής της υποεπιτροπής. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον πρέσβη Σκόγκ για την πλούσια παρουσίασή του, η οποία δεν μπορούσε παρά να είναι πλούσια λόγω ακριβώς της εξαιρετικής προσπάθειας της οποίας έχει κάνει η Σουηδική Προεδρία και ο ίδιος ο πρέσβης Κόγκ. Τα θέματα τα οποία αντιμετώπισε είναι πάρα πολλά. Δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα να τα σχολιάσω όλα. Θα ήθελα όμως να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Ίσως τα πιο ενδιαφέροντα από τα σημεία τα οποία παρουσίασε ο κύριος Πρέσβης. Να ξεκινήσω σχετικά με την διαθεσιμότητα εκπαίδευσης προσωπικού για τις πολιτικής μορφής παρεμβάσεις, όχι τις στρατιωτικές παρεμβάσεις μας και δράσεις μας. Εγώ συμμερίζομαι, θα έλεγα, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σκόγκ ότι από τη μία δηλαδή πρόκειται για μια εθνική ευθύνη των χωρών δηλαδή που συνεισφέρουν σε προσωπικό. Από την άλλη όμως, καλό θα ήταν να κάνουμε κάτι περισσότερο σε επίπεδο των πλέον βέλτιστων πρακτικών για να λειτουργήσουμε, για να λειτουργήσουμε ε, προς την κατεύθυνση πιο ομοιογενών ε, μηχανισμών και να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τα προφίλ των ανθρώπων που θα είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο που μέσω ακριβώς της σύγκλησης των μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του προσωπικού θα είναι ιδιαίτερα εύχριστα για τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ομοιογενοποίηση των συστημάτων κατάρτισης του προσωπικού που χρησιμοποιείται στις εξωτερικές δράσεις. Ένα άλλο ερώτημα αφορά το πώς έχει προχωρήσει η συζήτηση, η κοινή συζήτηση στο Συμβούλιο για την αποστολή Αταλάντα, για την δράση Αταλάντα. Αυτή η παρακολούθηση σαν παράδειγμα των αλλιευτικών δραστηριοτήτων η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό. Αυτό είναι ένα θέμα θα έλεγα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί, είναι ένα θέμα περίπλοκο. γιατί ο ευρωπαϊκός αλλιευτικός τόλος είναι πάρα πολύ συχνά θύματα των πειρατικών δραστηριοτήτων και ήταν εκτός ορίων ουσιαστικά μέχρι τώρα της αποστολής της συγκεκριμένης, της αποστολής Αταλάντα, τώρα όμως έχει συμπεριληφθεί στις δραστηριότητές της, όπως ε, έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα βοηθήσει και την καταπολέμηση των παράνομων αλλιευτικών δραστηριοτήτων, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε καλύτερα τις ανάγκες των νόμιμων Ευρωπαίων αλλιέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες με λίγα λόγια γύρω από τον τρόπο που εξελίσσεται η συγκεκριμένη δράση, η δράση Αταλάντα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις τώρα. Διάβασα μία δήλωση για την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει μία συναλλικότερη αντιμετώπιση του αφγανικού προβλήματος. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να καταλάβω καλύτερα εδώ τι εννοείται. Το πρόγραμμα δράσης, το Action Plan για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν είναι κάτι το ιδιαίτερα φιλόδοξο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάτι το πολύ σημαντικό, κάτι όμως το οποίο δια... λειτουργεί θα έλεγα με πολύ διάσπαρτο τρόπο και δείχνει ότι υπάρχει μια ουσιαστική έλλειψη κάποιων συνθετικών προσπαθειών, συνθετικών μέσων για την βελτιστοποίηση της ευρωπαϊκής παρέμβασης στην περιοχή. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα βήματα, αν έχουν αναλυφθεί συγκεκριμένα βήματα για τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος δράσης. Και σε ποιο βαθμό ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να μας βοηθήσει να αναπροσδιορίσουμε το προφίλ της συγκεκριμένη αποστολής και πά στο Αφγανιστάν. Σε το ότι είναι βέβαια δύσκολη η αποστολή, υπάρχει ένα θέμα αύξηση των αριθμών, αλλά δεν είναι εκεί αν θέλετε το πρόβλημα. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα ευχέρεια για το Αφγανιστάν. Αλλά θα ήθελα να μου πει ο πρέσβης Κόγκ λίγο περισσότερα πράγματα για τις προσπάθειες αποκατάστασης ε, της κρατικής λειτουργίας και ιδιαίτερα της κρατικής δικαιοσύνης στο Αφγανιστάν. Μία τελευταία παρατήρηση και κλείνω. Αναφερθήκατε σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο που αφορά την ε, προετοιμασία των δράσεων, το λεγόμενο Startup Fund. Αυτό εννοείται το Startup Fund, το, το Ταμείο Εκκίνησης Δραστηριότητας ή, ή σκοπεύετε να προτείνετε τη δημιουργία μιας νέας γραμμής στον προϋπολογισμό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεκδικεί ένα μείζωνα ρόλο σε σχέση με την λειτουργία αυτού του Ταμείου Εκκίνησης, του Startup Fund. Thank Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πράγματι δεν υπάρχουν ε, πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρόλα αυτά λίγοι έχουν παραμείνει εδώ. Να επανέλθω στο του Αφγανιστάν. Αναφερθήκατε στην παρουσία των αστυνομικών και είπατε ότι έχετε μόνο 100 ενώ θα θέλατε 400. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες ε, για τους ε, στρατιωτικούς μας ε, στο Αφγανιστάν. Δεν έχουμε διασφαλίσει την ασφαλειά τους, έχουμε θύματα και εφόσον δεν διασφαλίσουμε την ασφάλεια του προσωπικού αυτού, ιδιαίτερα των μη στρατιωτών, είναι δύσκολο να βρούμε ανθρώπους που να θέλουν να πάνε στο Αφγανιστάν. Thank you. Ευχαριστώ στον Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Προεδρία για την περιγραφή της πρόοδου. Και διακρίνω μια αισιόδοξη νότα. η οποία είναι και δέουσα σε μια στιγμή όπου η συνθήκη έχει τεθεί σε εφαρμογή, έχουμε γυρίσει πλέον μια σελίδα και έχουμε θέσει το πλαίσιο πλέον στη συνθήκη για την ε, γοργή αύξηση και ανάπτυξη της πολιτικής άμυνας και την δημιουργία μιας βασικής ομάδας για μια εταιρική συνεργασία. Θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις. να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να διατηρήσουμε τον τρόπο ζωής μας, τον πολιτισμό μας. από το τουβαλού. Αν ληφθούν οι κατάλληλες από το στρατιωτικό σκέλος της γραμματείας στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και έχετε την ε, εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη σκοπεύουν να αποστείλουν δημοσίους υπαλλήλου από τα Υπουργεία Εξωτερικών σε αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και ποιοτικό δηλαδή προσωπικό αλλά και επαρκές προσωπικό σε αριθμό. Κατά δεύτερον, πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός σχηματισμός του Συμβουλίου για τους ε, διαφόρους υπουργούς. Αυτό θα μπορούσαμε να το θέσουμε. Νομίζω ότι είναι ένα καλό θέμα. Μπορούμε να το θέσουμε τώρα Και τρίτη και τελευταία ερώτηση για το EGI. Μιλήσατε για ένα σχέδιο ενίσχυσης του. Θα ήθελα να ακούσω πιο πολλές ε, πληροφορίες, γιατί ο οργανισμός ενισχύεται βάσει της συνθήκης αν θα μπορούσαμε να αποδείξουμε στα Υπουργεία Εξωτερικών ε, Οικονομικών ότι πρόκειται για το πρώτο πρακτικό παράδειγμα μεγαλύτερης οικονομικής αποδοτικότητας εξαιτίας και χάρη στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι τότε θα έχουμε πετύχει ένα σημαντικό πολιτικό επίτευγμα. Και ένα τέτοιο πρακτικό πρώτο βήμα θα μπορούσε, αν θέλετε, να έχει αντίκτυπο και σε άλλους ε, τομείς δαπανών. Άρα θέλουμε διακαώς να στεφθεί με επιτυχία και να αποδείξει την αξία του στο κοινό το EGA. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρεσβευτή, να κάνω μια παρατήρηση και να θέσω και ερωτήσεις για το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν, το θέμα της ε, αύξησης των αστυνομικών δυνάμεων το έθιξε ο προηγούμενος ομιλητής. Όλοι ξέρουμε ότι 3 έως 4 χιλιάδες εκπαιδευτές αστυνομικοί χρειάζονται προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο αυτό εκπαίδευσης, αστυνομικής εκπαίδευσης, το οποίο είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα στην Ήπιθρο, προκειμένου να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση. Και τώρα, στα τέλη της Προεδρίας αυτής, διαπιστώνουμε εκ νέου ότι δεν έχουμε πετύχει τους στόχους που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς μπορούμε εμείς οι Ευρωπαίοι να προσμετρήσουμε την ε, σοβαρότητα και την αξιοπιστία της πολιτικής μας δράσης, της εξωτερικής πολιτικής μας δράσης. Μιλάμε για διάφορες αποστολές, αλλά σε μια τόσο σημαντική και θεμελιώδη σημασία αποστολή δεν ε, καταφέρουμε να υπερβούμε τα εμπόδια και να κάνουμε τη διαφορά, αν θέλετε. Σας ρωτώ λοιπόν πώς μετά από έξι μήνες εμπειρίας με το θέμα αυτό, πώς μπορείτε να αντιληφθείτε, πώς μπορείτε να φανταστείτε την πιο σοβαρή δραστηριοποίηση της Ευρώπης στο θέμα αυτό. Να μην συνεχίσει αυτή η επιφανειακότητα σε ό,τι αφορά την επιδίωξη των στόχων που εμείς ήδη έχουμε θέσει. Πέρα από το γεγονός ότι πάλι σε εμάς θα επανέλθει μπούμερανγκ το θέμα αυτό αν δεν τα καταφέρουμε. Δεύτερη ερώτηση αναφορικά με τη Σομαλία. Καταρχάς για την Αταλάντα. Το Κοινοβούλιο σε ψήφισμα έθεσε προς δύο τροποποιήσεις. Καταρχάς σε ό,τι αφορά τους αλληλείς και κατά δεύτερον την γεωγραφική επέκταση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε με ποιο τρόπο θα συμμετάσχει και το θέμα της αλληλείας και τι έχει να πει το Συμβούλιο για το θέμα της γεωγραφικής επέκτασης. Και κατά τρίτον, το Κοινοβούλιο υπέδειξε επίσης ότι η παράνομη αλληλεία και η παράνομη συσσόρευση αποβλήτων ε, στη Σομαλία αποτελούν θέματα τα οποία θα πιστούν και θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς το Συμβούλιο σκοπεύει να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες της σε ό,τι αφορά την αποστολή εκπαίδευσης. Ποια κράτη έχουν επιδείξει ως τώρα ενδιαφέρον ή ενδεχομένως να έχουν εκδηλώσει και προθυμία για να συμμετάσχουν σε τέτοιες αποστολές. Η Σομαλική Υπηρεσιακή Κυβέρνηση έχει επισήμως ε, υποβάλει αίτημα για τέτοια ε, αποστολή ή έχει εκφραστεί θετικά. Η έκθεση του ΟΗΕ του Νοεμβρίου έχει απαιτήσει ή έχει ενθαρρύνει, εν πάση περιπτώσει, τέτοια αποστολή εκπαιδευτική. Το Συμβούλιο ήξερε ότι ο πρόεδρος Σαρίφ απείλησε τους νέοεκπαιδευόμενους στρατιωτικούς ε, ε, στρατιώτες με επιβολή του νόμου της Σαρία σε περίπτωση που πουλούσαν όπλα. Βοηθάει αυτό στην όλη κατάσταση. Και τέλος, έχει σημειώσει το Συμβούλιο το γεγονός ότι ο ΙΕ υπέδειξε ότι η Σομαλία για το 2010 επαπειλείται με ανθρωπιστική κρίση ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα μέσα και αποτελεί πραγματικά προτεραιότητά μας να χορηγούμε χρήματα για μια τέτοια αμφιλεγόμενη αποστολή ή μήπως θα ήταν πιο μεγάλη προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ενδεχόμενη ανθρωπιστική κρίση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κόβαλ. E, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη, πρέπει να φύγω πολύ σύντομα. Θα ήθελα όμως να σας θέσω ένα ερώτημα. Ε, ε, οι συνεργάτες μου θα σημειώσουν την απάντηση. Άκουσα σήμερα τον Υπουργό Μπίλτ και άκουσα και εσάς και με ικανοποίηση διαπιστώνω τον τρόπο που εργάστηκε η Σουηδική Προεδρία και δεν νομίζω ότι μόνο εγώ το πιστεύω αυτό. Έχω μια ερώτηση για το Αφγανιστάν που αφορά και τις εκλογές και την ε, αλλαγή στην κοινωνία του Αφγανιστάν. Η ερώτησή μου είναι, οι πολιτικές προσπάθειες εκεί, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, προς ποια κατεύθυνση κινούνται, ποια συγκεκριμένα μέτρα χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες στην κοινωνία, οι οποίες ε, να διασφαλίσουν ε, το στόχο μας. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε τη γνώμη μου, αλλά εγώ διαπιστώνω ότι πολύ λίγο ε, συζητιέται το θέμα και ε, πολύ περιοριστικά θα ήθελα τη θέση σας ε, με βάση τις εμπειρίες σας των τελευταίων μηνών. Ευχαριστώ, Λούζιν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη, για την παρουσίασή σας. Επιτρέψτε μου να πω ότι βρήκα κάπως θολή την παρουσίασή σας ε, και δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις θέσεις σας. Ε, μιλήσατε για επιτυχίες. Ποιες επιτυχίες? Με ποιους στόχους μετράτε τους ε, στόχους σας. Είπατε ότι διαμεσολαβήσατε μεταξύ πολλών μερών. Ποιων μερών, ποιες, ποια βήματα πρόοδου επετέχθησαν. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπιτικόφερ. Σομαλία. Ποιο είναι ο στόχο σα στη Σομαλία? Είπατε ότι ένας στόχος είναι να ε, σταθεροποιηθεί η μεταβατική κυβέρνηση και η μεταβατική αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τη στήριξη του λαού, δεν είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένη, είναι διεφθαρμένη και η πολιτική της ε, είναι αμφιλεγόμενη. Ε, η Σαρία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, εφαρμόζεται όλο και περισσότερο, εφαρμόζεται κατά των γυναικών, είχαμε λιθοβολισμούς γυναικών. Αυτό είναι ο στόχος μιας ε, αποστολής εκπαίδευσης, να υποστηρίξει μια τέτοια κυβέρνηση. Θα μπορούσε να αποψιαστεί κανείς ότι υπάρχουν άλλοι στόχοι στη Σομαλία, οι οποίοι δεν, δεν ε, σαφείς. Ποιοι είναι οι στόχοι σας στη Σομαλία και τι μπορεί να επιτευχθεί ώστε να μπορείτε εκ των υστέρων να μιλάτε για επιτυχία όσον αφορά την αποστολή. Δεύτερη ερώτηση. Είπατε ότι θέλετε μια καλή εξωτερική υπηρεσία. Τι εννοείτε με αυτό για μένα. Μια τέτοια υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί δημοκρατικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η, Σουηδική Προεδρία όμως μιλά για μια τέτοια υπηρεσία ανεξάρτητη από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και στην περίπτωση αυτή ε, το δικαίωμα ε, ε, συναπόφασης του Κοινοβουλίου τι μορφή θα έχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζέμκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις παρατηρήσεις έχω. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ την Σουηδική Προεδρία. Θεωρώ ότι πράγματι επιτεύχθησαν πολλά βήματα προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Αυτό που χαρακτηρίζει την Σουηδική Προεδρία μεταξύ άλλων είναι ότι ε, έχουν εφαρμόσει πιο ρεαλιστική πολιτική. Μπορεί κανείς ε, να λέει πολλά, αλλά σημασία έχουν οι πράξεις ε, και το επικροτώ αυτό. Δύο σημαντικά πράγματα θα ήθελα να πω. Καταρχήν, συμφωνώ με τον κύριο Πρέσβη όσον αφορά την εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά τους σχηματισμούς μάχης. λέτε ότι θα συμβάλλετε στην ασφάλεια, δεν υπάρχει όμως κανένα πρακτικό παράδειγμα ε, όπου ε, ένας τέτοιος σχηματισμός έχει συμβάλει στην ειρήνη. Είτε θα έχουμε σχηματισμούς οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται ή ε, όλα είναι απλά ένα γραφειοκρατικό τέρας που δεν ωφελεί κανέναν. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο αυτό για την ε, αυτοπεποίθηση κάποιου, όχι όμως για την ασφάλεια. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να συνεχίσουμε ε, να κάνουμε σαν να μην υπάρχει πρόβλημα με τους σχηματισμούς τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούνται καν. Το Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν προφανώς οι ανθρωπιστικές προσπάθειε θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ε, μέτρα δηλαδή που βελτιώνουν ε, τις συνθήκες για το, τους πολίτες. Και ο αγώνας στο Αφγανιστάν ε, θα πρέπει να γίνει ε, μαζί με τους Αφγανούς. Αν δεν, ε, αν δεν στηρίζει ο λαός την κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα για το λαό. Και η ανθρωπιστική βοήθεια απαιτεί όχι μόνο χρήματα, εσείς θα διαθέσετε ένα δισεκατομμύριο, χρειάζεται όμως και ένας πολύπλοκος γραφειοκρατικός μηχανισμός. Αυτό συχνά ξεχνιέται. Και στην περίπτωση του Αφγανιστάν ναι, αυτό είναι δυνατό μόνο με τη συμμετοχή κάποιων χωρών. Για παράδειγμα, η Ρωσία και η Κίνα θα πρέπει να συμμετάσχουν και αυτές. Στις ανθρωπιστικές προσπάθειες ε, στο Αφγανιστάν ε, θα πρέπει ε, όσον αφορά τα θέματα επιμελητίας και τις μεταφορές να συμμετάσχουν τουλάχιστον η Ρωσία και η Κίνα. Επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πάρα πολύ για ο κύριος Πρέσβης, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για τις ε, σκέψεις που ακούσαμε. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχήν όσον αφορά το προσωπικό από την πολιτική πλευρά, από την πλευρά των πολιτών. Όπως είπατε κυρία Γκουαλτιέρη, πράγματι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν το προσωπικό. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει Έχουμε πετύχει πρόοδο στο σημείο αυτό, έχουμε συγκεντρώσει το δυναμικό μας ε, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο και ε, ενιαίο επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό κάναμε δηλαδή, συγκεντρώσαμε τις ομάδες μας ε, στις ομάδες αντίδρασης για τις κρίσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Γεωργίας όπου στείλαμε μια τέτοια ομάδα πριν ε, οργανωθεί επίσημη αποστολή. Η συγκέντρωση του δυναμικού μας ε, που, ώστε να μπορούν εμπειρογνώμονες να ασταλούν ε, πολύ σύντομα σε κάποιες χώρες θα είναι πολύ καλή, όπως έγινε άλλωστε στην περίπτωση της Γεωργίας. Όσον αφορά την αλία, αυτό το ανέφεραν αρκετοί. Η κατάσταση έχει ως εξής. Η εντολή Δεν το καλύπτει αυτό ρητά και απαντώ και στην κυρία Λουίζινγκ. Η ε, αποστολή στην Αταλάντα είναι ανθρωπιστικής φύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει με στρατιωτικά μέσα προσπαθώντας να βοηθήσει τον ε, λαό της Σομαλίας μέσω της ε, επιχείρησης Αταλάντα. και είχαμε 100% επιτυχία με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων. Δεν είχαμε ούτε μία απώλεια ε, από τότε που ξεκίνησε η αποστολή αυτή πριν ένα χρόνο. Όλοι λοιπόν ε, συμμετέχουμε. Εγώ προσωπικά Πήγα και θα ήθελα να ενθαρρύνω και εσάς να πάτε, ε, να δείτε την αποστολή. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί μερικές φορές ε, συναντούν άλλες παράνομες δραστηριότητες, ε, εμπορία ανθρώπων, ε, λαθρεμπόριο όπλων και κάνουν ε, ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις και να αναφέρουν τα περιστατικά. Υποθέτω ότι εάν συναντούσαν περιστατικά λαθρέας αλληλείας θα χρησιμοποιούσαν τα συστήματα που έχουν για να ενημερώσουν τις αρχές. Στην εντολή όμως όσα έχει αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται. Θέλουμε να κάνουμε την ανθρωπιστική δουλειά και να βοηθήσουμε την ε, κανονική ναυτιλία που συμπεριλαμβάνει την ε, νόμιμη αλληλεία. Αλλά από την πολιτική πλευρά και εδώ αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε το δυναμικό. Δεν νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλες τις φρεγάτες ε, και τις, ε, ε, τα στρατιωτικά μέσα που θέλουμε να κινητοποιήσουμε το 2010. θα πρέπει λοιπόν για την επιχείρηση αυτή να φροντίσουμε να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και το κατάλληλο δυναμικό, το κατάλληλο προσωπικό. Εντύπωση που είχαμε Η εντύπωση που λάβαμε όταν ε, φτάσαμε εκεί ήταν ότι οι ε, αεροπορικές περιπολίες ήταν πολύ σημαντικές και αποτελεσματικές, διότι με την ε, σημερινή τεχνολογία μπορεί κανείς να καλύψει μια τεράστια περιοχή. Μιλάμε για περιοχή που έχει το μέγεθος της Ευρώπης. Μπορεί λοιπόν να παρακολουθήσει κανείς από αέρος τι γίνεται πάνω σε μεμονωμένα πλοία. Είτε μιλάμε για πειρατικά πλοία, είτε για πλοία ε, τα, ε, τα οποία αποτελούν βάση για άλλες ε, παράνομες δραστηριότητες. Για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Και ιδιαίτερα το Αφγανιστάν που αναφέρατε πολλοί από εσά. Καταρχήν, ε, όσον αφορά... Όσον αφορά την EU4, στην απόφαση αναφέρεται ο αριθμός 400. Στην αρχή είχαμε πει 200, ε, τώρα μιλάμε για 400. Ε, θα πρέπει όμως ε, να μάθουμε από αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το κατάλληλο πρότυπο για το μέλλον. Είναι σημαντικό να αποφασίσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε και να προσαρμόσουμε τους αριθμούς ανάλογα. Αυτό είναι το ένα μάθημα που θα πρέπει να μάθουμε. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αποστολέ εάν δεν βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ετοιμότητα από πλευρά των κρατών μελών για κινητοποίηση. Και αυτή είναι η συζήτηση που είχαμε και στην περίπτωση τη Σομαλίας. Ενώ σχεδιάζουμε την επόμενη αποστολή, ε, εκπονούμε και ένα κατάλογο σχετικά με το ποιε χώρε είναι διατεθειμένε να συμμετέσχουν στι αποστολέ αυτέ. Ε, κάποιοι με ρώτησαν για ποιε χώρε μιλάμε. Ε, αρκετά κράτη-μέλη πήραν πρωτοβουλία. Η Ισπανία έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο. Η Γαλλία δραστηριοποιείται στο Τσιμπουτί με την αποστολή τη εκεί και υπάρχουν και άλλα κράτα-μέλη. Δεν έχω μπροστά μου τον κατάλογο. Ε, ας μιλήσουν μόνο τους τα κράτη-μέλη αυτά που έχουν ε, ε, δηλώσει την ε, ετοιμότητά τους και τη διάθεσή τους ναι, να συμμετάσχουν σε σχετική αποστολή. Αυτά για την UPOL. να επανέλθουμε στο Αφγανιστάν όμως. Ο στόχος της UPOL δεν είναι να αστυνομεύει όλο το Αφγανιστάν στόχος της ε, αποστολής αυτής ε, και εδώ διαφέρει από άλλες επιχειρήσεις ε, του ΝΑΤΟ και άλλων κρατών μελών. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν είναι ότι εργαζόμαστε σε στρατηγικό επίπεδο, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον Υπουργό, ώστε να παρέχουμε στρατηγικές συμβουλές σχετικά με το πώς οι ίδιοι Αφγανοί καλό θα ήταν να να αλλάξουν τις αστυνομικές τους δυνάμεις, να μεταρρυθμίσουν τις αστυνομικές τους δυνάμεις. Ε, δεν έχουμε πετύχει ακόμα πολύ καλά αποτέλεσματα όπως ξέρετε. Υπάρχουν όμως και άλλες προκλήσεις τις οποίες θα ήθελα να αναφέρω διότι ε, με ρωτήσατε σχετικά. Το γεγονός ότι δεν έχουμε συμβατική σχέση ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αυτό αποτελεί πρόβλημα. Κάποιοι αναφέρθηκαν σε κάποιες πτυχέ της EUPOL ε, και μία από τις δυσκολίες ε, κατά την προσέλκυση αστυνομικών στην EUPOL είναι ακριβώς αυτή. Θα πρέπει να έχουμε συμφωνία με την ISAF όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία και ε, πολλοί συμμετέχουν στα λεγόμενα PRT σε όλη την ε, χώρα ε, και αυτά θα πρέπει να συνεργάζονται με την αστυνομική αποστολή και αυτό θα πρέπει να γίνει με συμβατικές διευθετήσεις, αλλά υπάρχει καθυστέρηση. Τρίτη παρατήρηση για την UPOL. Το θέμα δεν είναι οι 320, αν δεν κάνω λάθος, αστυνομικοί ε, που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε προσθέσει 100 ε, επί Σουηδικής Προεδρίας, δηλαδή είμαστε πάνω, ε, έχουμε ξεπεράσει τους 300. Στόχος τους πάντως είναι να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν έχουν στόχο να εκπαιδεύσουν τον κάθε αστυνομικό του Αφγανιστάν. Στόχος τους είναι να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές των αστυνομικών. όσον αφορά τις προκλήσεις του Αφγανιστάν με τις οποίες ανέφερε και ο Κάρλ Μπίλτ. Κάποιες λέξεις κλειδιά, συγγνώμη αν είμαι ασαφής. Η αίσθηση ιδιοκτησίας ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο σαφείς απέναντι στις ε, αφγανικές αρχές. Είναι δική τους χώρα για να τους ε, βοηθήσουμε θα πρέπει να υπάρχει πολύ περισσότερη λογοδοσία όσον αφορά τη διαφθορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, αξίες που αντιπροσωπεύουμε. Πολύ συχνά οι Αφγανοί μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συνεπής. Όταν μιλάμε με μία φωνή το λέμε, αλλά τα μεμονωμένα κράτη-μέλη ε, συνεργάζονται με ε, ε, ε δημάρχους και άλλους συνομιλητές στη χώρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς, να αρνούμαστε, να έχουμε συναλλαγές με ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι διεφθαρμένοι. Και Γι' αυτό προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωση που εν μέρη θα αντικαταστήσει τις διμερεί πολιτικές που ε, είχαν κάποιες χώρε. Με καλύτερο συντονισμό δηλαδή θα μπορέσουμε να είμαστε και πιο ισχυροί ε, όταν επιμένουμε στην ε, λογοδοσία, στην καταπολέμηση της διαφθοράς κτλ. απέναντι στου Αφγανού. Άλλη σημαντική πτυχή εδώ είναι ο συντονισμός δεν ε, έχουμε συντονιστεί με τη διεθνή κοινότητα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι τεράστια δύναμη και ε, εάν κάποιο είναι μεγάλο, ε, δεσπόζει και στη συζήτηση μεταξύ άλλων και όσον αφορά τι πολιτικέ που αφορούν το Αφγανιστάν. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε στενή συνεργασία και συνομιλίε με του Αμερικανού και θα έχουμε πολύ περισσότερη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη, διότι έτσι ε, θα γίνουμε κατάλληλο συνομιλητής για τους Αμερικανούς. Πιστεύω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε κάποιο βαθμό. Το τρίτο θέμα εδώ είναι να ενισχύσουμε τον ΟΗΕ, διότι εκπροσωπεί όχι μόνο τις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόκειται για μια ομπρέλα που καλύπτει και την Κίνα, τη Ρωσία, το Τατζικιστάν, το Πακιστάν, την Ινδία, όλους αυτούς τους διεθνείς παράγοντες ε, θα τους καλύπτει λοιπόν μία ομπρέλα όπου υπάρχει και ε, νομοποίηση του ηγετικού ρόλου της. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το θυμόμαστε στην ε, μελλοντική μας δουλειά. Όσον αφορά την χρηματοδότηση πολιτικών αποστολών, στόχος μας δεν είναι... Δεν είναι αυτός ο στόχος του Startup Fund. αυτό θα δημιουργηθεί με τη νέα συνθήκη και θα καλύπτει στρατιωτικές αποστολές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει σημαντικό ρόλο εδώ. Αλλά στη σχετική γραμμή του προϋπολογισμού σημαντικό είναι να φροντίσουμε να υπάρχει περιθώριο για γρήγορη κινητοποίηση πολιτικών αποστολών. Δεν μιλάμε για πολλά χρήματα, θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να μην υπάρχει καθυστέρηση όταν υπάρχει ανάγκη για κινητοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, λόγους προϋπολογισμού. Ε, ο κύριος Στάφ και άλλοι αναφέρθηκαν ε, ε, στο EDS και θα Και αναφέρομαι στον σκελετό που έχει προκύψει από τις ε, θέσεις των κρατών μελών, ε, των οποίων θα πρέπει να ε, γεμίσει, να το πω έτσι, η Κάθριν Άστον. Όσον αφορά το EDA, συμφωνώ. Κάποιοι θα, θεωρού, θα θεωρήσουν ότι έχουμε περιορίσει τη σημασία του με καθυστέρηση της τριετούς προϋπολογιστικής προοπτικής αλλά με τον προϋπολογισμό μπορεί να αναγκάσει κανείς έναν οργανισμό να επικεντρωθεί ε, σε, ε, σε λίγες δραστηριότητες. Νομίζω ότι το ίδιο e έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ε, ότι επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε κάποια σημαντικά θέματα και αποδεικνύουν τη σημασία τους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί καλή πλατφόρμα για το EDA. Νομίζω ότι απάντησα στα περισσότερα που ρωτήθηκαν για τη Σομαλία. Η κυβέρνηση ε, η μεταβατική κυβέρνηση είπε ότι θέλει την υποστήριξή μας. Δεν προέκυψε από το πουθενά η μεταβατική αυτή κυβέρνηση. Είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας ε, να διαμεσολαβήσει ώστε να βρεθεί μια λύση. Ελπίζω να μην διαφωνούμε σε αυτό. Μπορείτε να πείτε ότι βρίσκεται υπό απειλή από τις ε, εξτρεμιστικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένου του Αλσεμπάπ. Εγώ... Η κυρία Λούισινγκ ε, νομίζω ότι προτείνει να αποσυρθούμε και να αφήσουμε τους ε, Σομαλούς να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό όσο καλύτερα μπορούν. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει ούτε τις γυναίκες, ούτε τα παιδιά, ούτε το λαό της ε, Σομαλίας. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό με τρόπο που να μην βλάψει κανέναν. Συμφώνω με αυτό και γι' αυτό ακριβώς είπα στην αρχή ότι αν αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε την οδό αυτή, είναι ζωτική σημασία το πώς θα πραγματοποιήσουμε την εκπαίδευση. Εάν όμως το κάνουμε αυτό, Ε, αυτή δεν θα έχει στόχο να προωθήσει αυτές τις ε, κακές πρακτικές που αναφέρατε, τους λιθοβολισμούς, ε, τη σαρία κλπ. Ε, θέλουμε να εξάγουμε ε, το καλό επίπεδο εκπαίδευσης ε, που γνωρίζουμε και στο οποίο είμαστε πάρα πολύ καλοί. Αλλά δεν ε, περιμένω να συμφωνήσετε. Πάντως αυτή είναι η θέση και των Ηνωμένων Εθνών και των Ηνωμένων Πολιτειών και των περισσότερων κρατών και ανθρώπων της περιοχής. Μαζί με άλλους έχουμε να παίξουμε ρόλο, όχι μόνοι μας. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να ενταχθεί στο γενικό πολιτικό πλαίσιο. Διαμεσολάβηση. Κυρία Λουίζινγκ, δεν είπα... Νομίζω ότι ο Καρλ ε, το ανέφερε, αλλά εγώ δεν είπα ότι ότι έχουμε μεσολαβήσει με επιτυχία. Αυτό που είπα ήταν ότι προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα, έναν μηχανισμό με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να μεσολαβεί καλύτερα. Έχουμε συχνά εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες περιοχές, στην Γεωργία, το κέρας της Αφρικής, το Σουδάν, το Αφγανιστάν. Αυτούς θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε στη δουλειά που κάνουν ε, όσον αφορά τη διαμεσολάβηση και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Θελήσαμε να βελτιώσουμε την υποστήριξη προς αυτούς τους ανθρώπους σε τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι απάντησα περισσότερο. Ο κύριο Νταφ ρώτησε σχετικά με του υπουργού αμήνη ή μάλλον για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και πώ σχετίζεται αυτό με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Δεν νομίζω ότι η συνθήκη προβλέπει ξεχωριστέ συναντήσει των Υπουργών Αμήνη. Μπορεί να είναι θέμα ερμηνεία και μπορεί η νομική υπηρεσία να έχει ε, γνώμη για το θέμα αυτό, αλλά Εμεί έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Πάντω ε, νομίζω ότι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εμεί κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα ήταν ε, να συμμετέχουν όσο γίνεται οι Υπουργοί Αμήνης ε, και υπάρχουν κάποιε πτυχέ, και νομίζω ότι αναφέρθηκατε σε κάποιε από Ε, Η δομημένη συνεργασία, η ρήτρα αλληλεγγύη είναι θέματα, ε, παραδείγματα θεμάτων όπου θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο οι Υπουργοί Αμήνης. στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή θα πρέπει να ε, συνεισφέρουν στα ε, Συμβούλια ε, Γενικών Υποθέσεων. Υπάρχουν γενικά θέματα όπου θα πρέπει οι Υπουργοί δεύτερου και τρίτου πυλών να συνεργάζονται στενά. Πάντως αυτέ οι συζητήσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Οι σχηματισμοί τα battle groups δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμή, ε, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι θα είναι ε, σημαντική συζήτηση αυτή. Νομίζω ωστόσο ότι μπορεί να ε, υποστηρίξει κανείς ότι δεν πρόκειται απλά για τέρας της γραφειοκρατίας. Ε, έχουν βοηθήσει πολύ τους Σουηδούς σε ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μας βοήθησαν να ε, μετατρέψουμε την εθνική μας άμυνα σε άμυνα που προσανατολίζεται πολύ περισσότερο σε διεθνείς συγκρούσεις και στους στρατιωτικούς κύκλους της Σουηδίας. Αναγνωρίζεται γενικά ότι η ασφάλεια πετυχαίνεται περισσότερο στο εξωτερικό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και σε κάποιες περιπτώσεις με τον ΝΑΤΟ επικεντρωνόμαστε στην ε, εδαφική μα άμυνα. Οι σχηματισμοί αυτοί λοιπόν ήταν πολύ χρήσιμοι για να, τη αυξήσουμε τη διαλειτουργικότητα. Συμφωνώ μαζί σας όμω, ότι το γεγονό ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ε, αποτελεί πρόβλημα αξιοπιστίας πιθανότατα, πολιτικό πρόβλημα δηλαδή, για το... Ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω ε, γι' αυτό ακριβώς επικροτούμε τη συζήτηση ε, επί του θέματος ε, για να γίνει αυτό ένα μέσο πιο φιλικό προς το χρήστη, να το πούμε έτσι, στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό στο συνάδελφο Μπίτι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου φτάνει το μισό λεπτό. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε, κύριε Πρεσβευτά, στην Αταλάντα και στην Αλία και είπατε δύο πράγματα. Καταρχάς ότι η προστασία της Αλλίας δεν αποτελεί ρητά τμήμα τη εντολής και κατά δεύτερον ότι οι αλλιευτικό στόλο θα, θα συνοδευτούν. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε, θα πρέπει να αλλάξει κάτι στην διατύπωση της εντολής, θα αλλάξουν τα πράγματα πρακτικά. Πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή. απάντηση. Σας ευχαριστώ. Δεν ήμουν πολύ σαφής ίσως για τον εξή λόγο. Συνεχίζονται ακόμα οι συζητήσει σε ό,τι αφορά την ε, εντολή, κατά πόσο θα γίνει α, τροποποίηση της εντολής, αναθεώρησή της. Και το τρίτο θέμα που εμπλέκεται είναι ασφαλώς το θέμα των πόρων. Δεν ξέρετε δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την ε, παρουσίαση του Ναβάρχου Χάτσον για την τεράστια έκταση των ε, δράσεών μας και των, τους περιορισμένους πόρους που έχουμε. Άρα θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από τους βασικούς μας στόχους που είναι η ανθρωπιστική προστασία και η εξασφάλιση ιδιαίτερα στον κόλφο του Άντεν όπου ακόμα πολλά έχουν να γίνουν. Αλλά αν θέλαμε να προσθέσουμε στην εντολή την παρατήρηση της λαθροαλληλίας και την ε, συνοδεία των λαθρέων αλληλευτικών σκαφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει και για το Αφγανιστάν ίσως. Έχουμε τους πόρους αυτούς και τα τοξικά απόβλητα αποτελούν και αυτό ένα θέμα. Αλλά όπως σας είπα, η αποστολή αυτή και μετά από συζητήσεις μου με τους παράγοντες επιτόπου προσπαθεί καθένα να κάνει ό,τι μπορεί εντός των ορίων της εντολής τους. Συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων εμπορίας ε, ανθρώπων όπου έχει υπάρξει παρέμβαση ε, και μάλιστα με τρόπο που δεν αναφέρεται ρητά στην εντολή. Με έναν, αν θέλετε, κανονικό ανθρωπιστικό τρόπο. Αλλά σημειώνουμε την θέση του Κοινοβουλίου για την Αλία και νομίζω ότι η συζήτηση για την εντολή και την αναθεώρηση της ενδεχομένω ε, θα συνεχιστεί πάντα εντό των περιορισμών που μας επιβάλλουν οι υφιστάμενοι πόροι. Μάλιστα, ο Πρόεδρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, πρέσβη για τις πληροφορίες αυτές και τις απαντήσεις που μας έδωσε. Ήταν μεγάλη μας τιμή που σας είχαμε μαζί μας σήμερα. Μία ε, άλλη πληροφορία για έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο 10 Ιανουαρίου για μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Τζαντζίν για την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Είναι η τελευταία συνεδρίασή μας για φέτος. Σας εύχομαι λοιπόν καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Ευχαριστώ.